Συνεχίζουμε λοιπόν με τη συνεδρία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Καλωσορίζω τον κύριο Λεμέτρη, Γενικό Διευθυντή για την Περιφερειακή Πολιτική και την Αστική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέρασαν πολλοί μήνες από την ε, τελευταία φορά που ήρθατε. Καλώς ήρθατε λοιπόν ξανά και έχετε το λόγο για μια αρχική παρουσίαση και στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο τα μέλη της Επιτροπής μας για ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις. Ανάλογο δηλαδή με αυτό που θα μας πείτε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Μιχαήλοβα, αξιότιμα μέλη. Πράγματι έχει περάσει αρκετός καιρός. Στο μεταξύ όμως ε, ερχόταν η Επίτροπος Κρέτσου αρκετά συχνά και ελπίζω να μην το θεωρήσατε παράληψη από μέρους μας που δεν ερχόμουν. Είναι η κατάλληλη στιγμή λοιπόν να κάνουμε έναν απολογισμό του παρελθόντος, του παρόντος και να δούμε πώς προετοιμάζουμε το μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ γρήγορα και με χρονολογική σειρά σε όλα αυτά. Νομίζω πως η περίοδος 2017-2013 είναι μια περίοδος που δεν πρέπει να ξεχνάμε, διότι μας δίνει τα περισσότερα στοιχεία βάσει τα οποία θα σχεδιάσουμε το μέλλον. Η λήξη της περίοδου 2017-2013 ολοκληρώνεται αρκετά ομαλά, πολύ περισσότερο από ό,τι προηγούμενες. Επίσης, θα κοιτάξουμε και την ε, τρέχουσα περίοδο για να δούμε πώς εξελίσσεται και θα κοιτάξουμε τις δαπάνες στο τέλος του 2015. Θα δούμε ότι παρά την ε, σοβαρή οικονομική κρίση, την ε, πιο μεγάλη που αντιμετώπισε η Ευρώπη από το δεκαετία του 30, είχαμε αρκετά καλά ποσοστά απορρόφησης. Τώρα, θα βασιστώ στην παρουσίασή μου σε αυτές τις ε, γραφικές παραστάσεις. Εδώ η πρώτη απεικονίζει την ταχύτητα υλοποίησης το 2014 και το 2020. Δεν θα σας εκπλήξει ότι το 2020 είχαμε χαμηλότερα ποσοστά. Και σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική υλοποίηση, Ω προ τι ενδιάμεσε πληρωμές, δηλαδή προς τα κράτη-μέλη, βλέπουμε ότι στο τέλος του 2018, δηλαδή στο τέλος του πέμπτου έτους του υφιστάμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, ήμασταν μόλις κάτω από το 2% ε, σε πληρωμές, δηλαδή έχουμε πολύ ακόμα. Τώρα, σε σχέση με το 2007-2013, που μην ξεχνάτε ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, διότι καλύπτει ε, το 2009 ως 2011, είχαμε πέντε ποσοστιαίες μονάδες ε, πιο πάνω. Ήμασταν πάνω από το 25% υλοποίηση. Παραμένουν λοιπόν αργά τα πράγματα και παρατηρούμε ότι δεν κλείνουν τα κενά και δεν μπορούμε να φτάσουμε στα νούμερα του 2007-2013. Τι συμβαίνει λοιπόν, γιατί όλα αυτά. Κάναμε έναν απολογισμό και είδαμε ότι κανείς δεν θα μας περιμένει, η ταχύτητα είναι βασική και η συνοχή έχει στόχο να στηρίξει τα κράτη-μέλη σε, σε αυτήν την ε, μεταβατική διαδικασία στην οποία βρίσκονται έχει άμεση σχέση με την ε, φιλοδοξία μας για έναν πλανήτη βιώσιμο, μακροπρόθεσμα, για τεχνολογική πρόοδο. Και δεν μπορούμε επομένω να λέμε πως ένα-δυο χρόνια δεν έχουν σημασία στο αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε σε αγώνα δρόμου με τις ΗΠΑ και με την Κίνα και χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι είναι κατάλληλη η διαδικασία, ότι μπορεί να στηρίξει εγκαίρως τα κράτη-μέλη για αυτήν την ε, μετάβαση στην οποία βρίσκονται. Από αυτή τη γραφική υπέσταση βλέπουμε ότι χρειάζεται περισσότερη δημοσιονομική πειθαρχία από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μια ανταλλαγή ανάμεσα στην ταχύτητα και στην ποιότητα των ε, δαπανών. Έτσι μας λένε. Αυτό όμως για μας δεν ισχύει. Αυτό που καταφέραμε στην περίοδο 2017-2013 με τον ΙΣΙΝ 2 είναι ότι είχαμε νέα κρατημέλη, περισσότερα ε, κονδύλια, λιγότερη εμπειρία. Και τι γίνεται 14 χρόνια αργότερα. Βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη αυτά τώρα έχουν συνηθίσει στην επιμερισμένη διαχείριση και στην εφαρμογή και υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Γιατί λοιπόν να είμαστε πιο ελαστικοί στο μέλλον, ενώ βλέπουμε ότι είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στο παρελθόν, χωρίς να είμαστε πιο ελαστικοί. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε με μεγαλύτερη προσοχή το, μεγα... το πιο προβληματικό σημείο, δηλαδή το πέρασμα από τη μία περίοδο στην άλλη. Παρατηρήσαμε ότι υπάρχει μία διακοπή μεταξύ των περιόδων και έχουμε δει ότι αν αρχίζεις κάτι σε μία περίοδο πρέπει να το τελειώσεις την ίδια περίοδο και μετά πάλι από την αρχή. Ξεκινάς από το μηδέν την επόμενη περίοδο. Αυτό που προτείνουμε για το μέλλον είναι περισσότερη ευελιξία σε προγράμματα που τρέχουν σε μία συγκεκριμένη περίοδο και δεν προλαβαίνουν να τελειώσουν. Τα προγράμματα αυτά λοιπόν εμείς προτείνουμε να μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο. Κάτι το οποίο θεωρούμε θα βοηθήσει πάρα πολύ και θα διασφαλίσει μια συνέχεια ως προς την υλοποίηση και την ε, στήριξη των προγραμμάτων συνοχής. Αλλά για να μπορέσουμε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή υλοποίηση προγραμμάτων και για να έχουμε ένα καλό ξεκίνημα, είναι σημαντικό τα προγράμματα να εγκρίνονται εγκαίρως και όχι όπως γίνεται τώρα, όπου βλέπουμε πως πάνω από τα μισά προγράμματα εγκρίνονται κατά το δεύτερο έτος της ε, περίοδου προγραμματισμού, δηλαδή στην περίπτωσή μας το 2015. Περνάμε τώρα στην προετοιμασία για το μέλλον. Βλέπετε και την ε, σχετική γραφική παράσταση. Έχει να κάνει με την επιλογή των ε, προγραμμάτων. Εδώ είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, όμως νομίζω πως ε, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην υλοποίηση, διότι αυτό είναι και το μέτρο σύγκρισης. Βλέπουμε τι αλλάζει. Περνάμε τώρα στην προετοιμασία. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την νομοθετική διαδικασία. Και να πω λοιπόν ότι έχουμε μεγάλο θαυμασμό στους συνεισηγητές σας, ιδιαίτερα για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, την κυρία Κρέλ δηλαδή και τον κύριο Νόβακοφ. Ιδιαίτερα προς την κυρία Κρέλ, η οποία εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά το ότι είναι άρρωστη. Κατάφερε λοιπόν να πραγματοποιηθούν συναντήσεις, τριμερείς διάλογοι, όσο το δυνατόν συχνότερα στο χρονικό διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μας και αυτό σε μια εποχή όπου δεν είναι τόσο συχνή αυτή πολιτική πολιτικοί διάλογοι. Και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εκτιμούμε λοιπόν ότι έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα και σίγουρα θα θέλαμε να είχαμε επιτύχει κάποια συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για κάποιο ή κάποια από τα μέρη του κανονισμού κοινών διατάξεων. Νομίζω πως δεν ήμασταν πολύ μακριά από αυτό. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους στόχους της πολιτικής και τον προγραμματισμό. Σε αυτό ακριβώς το σκέλος χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να κινήσουμε τους ε, διαλόγους ανάμεσα στα κρατημέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μελλοντικά προγράμματα. Έχουμε λοιπόν μια κάποια λύπη για το ότι δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τα όσα είχαμε προγραμματίσει, όμως θεωρούμε πως ε, έγινε πολύ σημαντική δουλειά, πως δεν θα χαθούν αυτοί οι κόποι και θα μπορέσουμε να βασιστούμε στα όσα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα για να συνεχίσουμε. με την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Θεωρούμε λοιπόν πως η συζήτηση έχει επιφέρει σαφήνεια στα πιο σημαντικά σημεία, στα επίμαχα σημεία. Βέβαια, εντάξει, οι λεπτομέρειες παραμένουν ανοιχτές προς συζήτηση. Βλέπουμε όμως ότι τα βασικά στοιχεία της ε, περίοδου προγραμματισμού του κανονισμού κοινών διατάξεων έχουν αρχίσει να αποκτούν μία μορφή. Εμείς λοιπόν θέλουμε να θεωρούμε το ποτήρι μισογεμάτο. και πως μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε μια ικανοποιητική βάση για περαιτέρω συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Τώρα πώς προχωρήσαμε, πώς προετοιμαστήκαμε. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε η μελλοντική πολιτική συνοχής να συνδέεται στενότερα με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και αυτό διότι πιστεύουμε ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε εργαστεί πολύ για να μην καταπιεί το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο την πολιτική συνοχή. Για μας είναι δύο ίσα προγράμματα. στο μεταξύ. Θα είχατε, φαντάζομαι, την ευκαιρία να διαβάσετε τις ε, εκθέσεις ε, για την κάθε χώρα που δημοσιεύσαμε στο τέλος του Φεβρουαρίου. Τώρα, ποιο είναι το νέο στοιχείο αυτών των εκθέσεων που συνδέονται μεταξύ τους. Τι του συνδέει λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την πολιτική συνοχή. Πρώτον, ενισχύθηκαν τα στοιχεία για τις ανάγκες που υπάρχουν σε επενδύσεις στα κράτη-μέλη. Όλες οι επενδυτικές ανάγκες, όχι μόνο εκείνες που ίσως στηριχθούν από την πολιτική συνοχή στο μέλλον. Έχουμε δηλαδή και τις δημόσιες επενδύσεις και τις ιδιωτικές επενδύσεις σε όλους τους πιθανούς τομείς. Έπειτα, δεύτερο νέο στοιχείο στις ε, εκθέσεις αναχώρα είναι ότι εκτός από τις ε, χώρες τις οποίες δεν χρειάζεται, δηλαδή όπως για τη δική μου για παράδειγμα, για το Λουξεμβούργο, υπάρχει ένα νέο τμήμα το οποίο αναλύει τις ε, περιφερειακές ε, διαφορές και τις τάσεις που επικρατούν. Εξετάσαμε λοιπόν κάποια κράτη-μέλη τα οποία χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια. Δηλαδή από μια περιφέρεια, πούμε, για παράδειγμα τα κράτη της Βαλτικής, που στατιστικά θεωρούνται μια περιφέρεια. Σε αυτήν την ε, περιοχή λοιπόν ξεπεράσαμε αυτήν ε, την ε, έννοια της μίας περιφέρειας και είδαμε τις σημαντικές, όπως διαπιστώσαμε, διαφορές από χώρα σε χώρα. και αυτό μας οδήγησε σε συγκεκριμένες προτάσεις και συστάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις, θεωρούμε πως έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια αρκετά στεγανή βάση έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ανάλυση των προτεραιοτήτων για την πολιτική συνοχής. Αυτό φαίνεται στο παράρτημα Δέλτα, που είναι γνωστό πλέον. Είναι ένα παράρτημα δύο-τριών σελίδων, είναι αρκετά συμπυκνωμένο, όπου αναφερόμαστε στη νέα δομή της πολιτικής, που φυσικά είναι αντικείμενο συμφωνία μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου, και τους νέους στόχους πολιτικής. Αυτά τα παραρτήματα λοιπόν ακολουθούν αυτή τη δομή που προτείναμε για το μέλλον. Και όπως βλέπετε από αυτόν εδώ τον πίνακα, εξετάσαμε και τις επιπτώσεις αυτών των ε, κανόνων για θεματική συγκέντρωση. Όπως γνωρίζετε, αυτοί οι κανόνες αφορούν τη θεματική συγκέντρωση για τα πιο αναπτυγμένα κρατημέλη και θα καταστήσουν δυνατό οι στόχοι πολιτικής να είναι πιο επικεντρωμένοι σε συγκεκριμένα πράγματα. Η θέση μας λοιπόν με βάση την ανάλυση που έχει γίνει είναι ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη όπως η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία, η Δανία και η Φιλανδία τα οποία έχουν μικρή στήριξη από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Βλέπουμε ότι τα νούμερα από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι περίπου 10 ευρώ κατά κεφαλή ανά έτος. Χρειάζεται λοιπόν να σκεφτούμε πραγματικά πόσο μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά με ένα τόσο μικρό ποσό. Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι θα αποκομίσουμε τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη και τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία σε εκείνα τα κράτη-μέλη, εστιάζοντας μέσω του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης αποκλειστικά στην ε, καινοτομία και στην ευφύ ανάπτυξη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μέσα σε αυτές τις δαπάνες δεν θα υπάρχουν ε, δαπάνες που θα ωφελήσουν το κλίμα, για παράδειγμα. Διότι σήμερα δεν έχουμε την αναγκαία τεχνολογία, ούτε καν κάποιες πολύ βασικές τεχνολογίες έτσι ώστε να επιτύχουμε τους ε, στόχους για το κλίμα. Μετά βλέπουμε ότι κάτω χώρες είναι εντό αγωγικών ε, μία κατηγορία από μόνες τους. Ζητήσαμε λοιπόν να εισαχθεί και αυτή η εδαφική διάσταση δεδομένη στις μεγάλες αστικοποίησεις στις κάτω χώρες. Και βλέπετε τώρα ότι για χώρες όπως η Αυστρία και η Γερμανία ένα στόχος πολιτικής τον οποίο δεν θα συμπεριλαμβάναμε είναι η συνδεσιμότητα. Διότι δεν θεωρούμε πως δεδομένη της ε, μέτρια στήριξης προς την Αυστρία και τη Γερμανία και δεδομένων των ε, διαθέσιμων πόρων και των ε, εθνικών προγραμμάτων, είτε αυτά έχουν να κάνουν για την ανάπτυξη ευρυζωνικότητας, είτε για τη σύνδεση μεταξύ πόλεων, θα, θα ήταν σωστό να αποτελούν στόχο πολιτικής. Καλύπτονται λοιπόν από το στόχο πολιτικής νούμερο 3. Για όλα τα υπόλοιπα, λέμε πως υπάρχουν προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να ε, αναφέρει η πολιτική συνοχής και είναι οι τομείς 1 ως 5. Θέλουμε να τονίσουμε ότι το παράρτημα Δέλτα καθορίζει την αφετηρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν θα εισέλθει σε διμερείς διαπραγματεύσεις για μελλοντικές συμφωνίες, εταιρική σχέση ή διάφορα προγράμματα. Σίγουρα δεν είναι εξαντλημένη αυτή η λίστα. Σίγουρα μπορεί να αλλάξει. Μπορούμε για παράδειγμα να δούμε ότι στη Γερμανία μπορείς να ξοδέψεις εκατομμύρια για ένα συγκεκριμένο στόχο πολιτικής. Ε, αυτό πιο πολύ υπάρχει για να δούμε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε ως προς τις προτεραιότητες. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό αποτελεί μία ισχυρή βάση και μία ισχυρή αφετηρία για αυτό που θεωρούμε μια ανταλλαγή απόψεων πολύ επικοδομητική με τα κράτη-μέλη σχετικά με, το, με τη μελλοντική μορφή των προγραμμάτων αυτών. Τέλος. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Αλλά πριν δούμε αυτό, να τονίσω ότι αυτό που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση με τις προτάσεις μας. είναι ο νομοθέτης να έρθει αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί να αποφύγει. Όλα αυτά λοιπόν με επιφύλαξη προς την νομοθετική διαδικασία, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να φτάσουν σε αυτή τη συμφωνία για τις λεπτομέρειες του κανονισμού κοινών διατάξεων, για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Και όταν θα συμφωνήσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τους κανόνες, θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το διμερή διάλογο έτσι ώστε να ολοκληρωθούν τα επιχειρησιακά προγράμματα με το κάθε κράτος μέλος. Βέβαια αυτά είναι εικασίες, αλλά πρέπει να τις κάνουμε έτσι ώστε να επιλέξουμε μία αφετηρία και αυτό γίνεται με το παράρτημα Δέλτα και την πρόταση της Επιτροπής. Δηλαδή είτε αυτό είναι θεματική συγκέντρωση, είτε έχει να κάνει με την επιλεξιμότητα ορισμένων δαπανών, ε, το, το εξετάζουμε από αυτήν την οπτική γωνία. Τα επόμενα βήματα λοιπόν έχουν ως εξής. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δούμε τι κεφάλαια υπάρχουν έτσι ώστε να κοιτάξουμε και τις ε, εκθέσεις ε, της κάθε χώρας ε, σε συνδυασμό με το παράρτημα Δέλτα και συνολικότερα την κατάσταση. Έχουν γίνει δύο συναντήσεις, μία στην Πράγα και μία στη Βαρσοβία και έμεινα ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την ανταπόκριση που είχαμε από τη συμμετοχή των φορέων σε αυτές τις δύο χώρες και από την ετοιμότητα που έδειξαν για να ξεκινήσουν τις διμερείς συζητήσεις. Για μας λοιπόν αυτές οι δύο χώρες ήταν ε, το η ήταν ιδανική περίπτωση για να δούμε πώς μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί με επιτυχία ένα τέτοιο πρόγραμμα. Καλέσαμε λοιπόν όλους τους ε, αρμόδιους φορείς να συμμετάσχουν και είχαμε μία πάρα πολύ καλή πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Τώρα σύντομα θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να μας δώσουν έναν οδικό χάρτη όπου θα αναφέρεται πώς εκείνα βλέπουν να διαγράφονται τα επόμενα βήματα έτσι ώστε να εγκρίνουν και επίσημα τα επιχειρησιακά προγράμματα μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Δεν θα υπάρξουν λοιπόν καθυστερήσεις σε αυτή την περίοδο. Και έχουμε προτείνει τα κράτη-μέλη να μας δώσουν τον οδικό χάρτη μέχρι τα μέσα του τρέχοντος έτους στη Βαρσοβία ήταν έτοιμοι, όπως σας είπα. Ήδη ήξεραν το χρονοδιάγραμμα, τι θέλαν, τους στόχους και είχαν την ίδια φιλοδοξία να τελειώσουν δηλαδή με την έγκριση μέχρι, τα, μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Τώρα, η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, όπως γνωρίζετε. Ακόμα υπάρχουν οι συστάσεις αναχώρα που πρέπει να υποβληθούν. Στις 5 Ιουνίου θα ε, δημοσιευτούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ έχουμε ακόμα κάτι καινούριο, μια σύνδεση, νέα σύνδεση με την πολιτική συνοχής και επίσης στις συστάσεις αναχώρα αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε επενδύσεις και επενδυτικές προτεραιότητες. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο φέτος. Δεν ξέρω αν θα σας εκπλήξουν αυτές οι συστάσεις, διότι είναι φυσική απόρρια των εκθέσεων αναχώρα. Σε αυτές τις συστάσεις για επενδύσεις δεν περιοριζόμαστε στην πολιτική συνοχής, αλλά στις γενικότερες επενδυτικές ανάγκες κάθε κράτους μέλους. Νομίζω πως μακρηγόρησα, αλλά αν υπάρχει χρόνος ε, θα ήθελα να ακούσω και τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και όχι καθόλου, καθόλου δεν μακρηγορήσατε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Φαίνεται ότι έχετε ένα σαφέ ε, σχέδιο κατά νου. Και το συζητήσαμε το πρωί. Συζητήσαμε το πρωί ποια είναι τα σχέδια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατά πάσα πιθανότητα τώρα θα έχουμε και ερωτήσεις. Οι συντονιστέ, φαντάζομαι. Ο κύριο Φάνι Τελρόι. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, ευκαιρία αυτή που μου δίνετε. Μεταξύ των δύο νομοθετικών αυτών περιόδων ε, είναι καλό να κάνουμε μια σύντομη παύση και να αναλογιστούμε. Μία ερώτηση λοιπόν έχω να κάνω. Μιλήσατε για το εξάμεινο, αλλά συμφωνήσατε και εδώ στην Επιτροπή αυτή επί του προγράμματος ε, υποστήριξη των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων και αυτό συνδέεται άμεσα με αυτά που συζητάμε γιατί περιλαμβάνει πολλές αλλαγέ. Πείτε μας λοιπόν πώς συνδέεται αυτά που μας λέτε για το εξάμεινο και με αυτά που μας είπατε για την εφαρμογή των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων γιατί νομίζω ότι μιλήσαμε για 70% περίπου των συστάσεων που συχνά συνδέονται με τις ε, συστάσεις ε, με την πολιτική συνοχή. Δεν άκουσα να το αναφέρετε όμως αυτό γιατί μιλάμε για μεγάλο χρηματικό ποσό, 20-25 δις την επόμενη προγραμματική περίοδο για διαδραστικές μεταρρυθμίσεις. Είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος, μήπως είναι η ίδια πλευρά του νομίσματος. Κατά δεύτερον, για την απόδοση δεν είπατε τίποτε. 25 δις ε, στις ε, εκθέσεις χώρα. Εγώ αναρωτιέμαι Τι γίνεται με αυτά τα 25 δισεκατομμύρια. γιατί ε, εμείς θέλουμε να υπάρχει να πάνε αλλά τι γίνεται αν περισσέψουν. Θα ήθελα να ξέρω την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Επίσης, είπατε ότι τα χρήματα από την περίοδο αυτή θα μεταφερθούν ε, κατευθείαν στην επόμενη περίοδο. Αυτό μην το πείτε όμως έτσι στους καθαρούς εισφορείς, γιατί θα σας πούν «Μα αφού δεν δαπανήθηκαν οι πορεία αυτοί, γιατί να τους ξαναβάλουμε στο ίδιο κορβανά». Νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο που θα πρέπει να πείτε. Γιατί αν το ακούσει αυτό ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών ε, δεν πρόκειται να μου στείλει ανθοδέσμη. τελευταία παρατηρήση. Συζητήσαμε για κάποια πράγματα τα οποία είναι στην εξουσία του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά πιλωτικές και προπαρασκευαστικές δράσεις. Ε, αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε στο παρελθόν για την ε, τοπική συνεργασία και την συνοχή. Έχουμε ειδικά προγράμματα τα οποία ξεκίνησαν από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ίσως θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την γραμματεία μας για να δούμε ποια πράγματα πάνε καλά και να μην περιμένουμε την ε, κρίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα τέλη της, Ευρωπα... περίοδου. Να το προκαταλάβουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ που ήλθατε εδώ, γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι μιλάμε για μεγάλα χρηματικά πόσα, παρά το γεγονό ότι υπάρχουν ε, και άλλα τμήματα πολλά χρήματα λοιπόν στο ERDF. Και άρα είναι ακόμα πιο σημαντικό. Εν και της μετακίνησης του πληθυσμού προς τις πιο πλούσιες χώρες. Υπογραμμίζω την αναγκαιότητα λοιπόν της εργασίας και τη δική σα και τη δική μα Σα ευχαριστώ. Γιατί μπορεί να μην σα είδαμε πολλέ φορέ, αλλά σα είχαμε συνέχεια στο μυαλό μα. Η πρόεδρο πολύ προσωπικό σχόλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Κρέλ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω τι εννοείται ακριβώ, κύριε Φανίστερο, με αυτή την τελευταία πρόταση, αλλά εν πάση περιπτώσει να το συζητήσουμε με ένα ποτήρι κρασί. Να σα ευχαριστήσω, κύριε Λεμέτρα, για την πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή που κάνετε στην Επιτροπή μας. Μία ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα. Είστε πολύ αισιόδοξο και χαίρομαι που ήδη μιλάτε με τους εταίρους και κάνετε προετοιμασία. Αλλά, ειλικρινά, πολύ αναρωτιέμαι κατά πόσο θα δικαιωθεί αυτή η αισιοδοξία. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το Συμβούλιο αποφάσισε περίπου 50% της πολιτικής συνοχής να μπει στο επόμενο πεδίο για το Πουδουπού. Έχετε ακούσει όλοι σας προφανώς ποια είναι η άποψη της Γερμανίας για τα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για το δεύτερο ημίση του 2020. Αν ληφθεί τότε η απόφαση για το 50% της πολιτικής συνοχής, δεν μπορώ να δω, να καταλάβω πώς θα την υλοποιήσουμε και νομίζω ότι έχουμε μέχρι τις 31 ε, ε, Δεκεμβρίου 2020 για τελικά αποτελέσματα. όπως και την προηγούμενη φορά έτσι έγινε. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει καθυστέρηση. Πιστεύετε ότι υπάρχει οποιαδήποτε δυνατότητα να ξεκινήσει ο προγραμματισμός πριν έχουμε στο τραπέζι μπροστά μας τον τελευταίο και τελικό κανονισμό κοινών διδάξεων. Δεν είμαι πραγματικά καθόλου σίγουρη για το πώς θα εκτελεχθεί η υπόθεση αυτή. Ίσως εσείς έχετε κάποιο παραπάνω στοιχείο και σχόλιο εκτός μικροφώνου του κυρίου Φανίστερο. Όχι, λέει η κυρία Κρέλ. Όχι, όχι, εγώ δεν ξέρω ποτέ τίποτα, λέει η κυρία Κρέλ. Αυτό επειδή είσαστε στην προεκλογική εκστρατεία, γι' αυτό δεν τα ξέρετε όλα. Όχι, όχι. Αυτό προφανώς και είναι αστείο. Λέει, πρόεδρος αστείευομαι. λίγο. Ο κύριος Φαμ Μίλτενμπουργκ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο Λεμέτρα για την ε, πολύ σαφή παρουσίαση και για την έκκληση για πιο μεγάλη δημοσιονομική πειθαρχία για τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτό το εκλαμβάνω και ως ε, έκκληση για αυτή η εφαρμογή του νησιν 2. Αλλά δυστυχώ ε, δεν έχουμε πάντα ό,τι θέλουμε. Το λέει και το τραγούδι. Μιλάω για την προπαρασκευαστική φάση για τη νέα προγραμματική περίοδο. Φυσικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε όσο πιο νωρίς γίνεται, αλλά εξαρτώμαστε και από τις διάφορες διαπραγματεύσεις για διάφορα νομοθετικά θέματα και εδώ δυστυχώς συμφωνώ με τους συναδέλφους μου που λένε ότι δεν σημειώσαμε επαρκή πρόοδο υπό την Ρουμανική Προεδρία. Δεν φταίτε εσείς φυσικά γι' αυτό. Πρέπει να επιταχύνουμε λοιπόν ως Κοινοβούλιο αυτό φυσικά τώρα θα είναι το καθήκον των νέων συναδέλφων στην Επιτροπή. Επίση, κάποιε ερωτήσει, γιατί υπήρχαν πολλά αμφιλεγόμενα θέματα στην Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη και η... του Ταμείου Συνοχή και η σχέση του με τα δίκτυα TNT, με το Connective Europe Facility. Ε, η συνεργασία πώς πάει τα τελευταία χρόνια με τους ε, συναδέλφους από την Γενική Διεύθυνση MOVE και πιστεύετε κι εσείς όπως και εγώ ότι αυτό έχει αποτελέσει επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Έχουμε απορροφήσει ουσιαστικά όλους τους πόρους στο ΣΕΦ από τα Ταμεία Συνοχής σε προγράμματα μεταφοράς, μεταφορών. Τι λέτε λοιπόν, να το συνεχίσουμε, μήπως έχετε κάποιες αμφιβολίες... Θα ήθελα μια ειλικρινή απάντηση. Ένα άλλο ακαθόδε θέμα αμφιλεγόμενο. Στον κανονισμό ERDF μιλήσατε για μη επιλέξιμες δραστηριότητε. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια συζήτηση και εγώ θα ζητήσω να τηρηθεί η γραμμή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τι ε, μη νόμιμες ε, αλλά θα υπάρξει μεγάλη συζήτηση. Για παράδειγμα, θα υπάρξει το θέμα των ρεκτών καυσίμων σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά αεροδρόμια, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, σιδηροδρομικέ μεταφορέ. Εγώ προσπαθώ να βρω και τα επιχειρήματα υπέρ και κατά. Μπορείτε να μα εξηγήσετε και να εξηγήσετε και στου συναδέλφου, εκ νέου γιατί η Επιτροπή θέλει να είναι πιο αυστηρή σε σχέση με τις ε, επιλέξιμες και μη δραστηριότητες. Τέλος. Το Μάιο του 2016 ξεκίνησε η ατζέντα για την Ήπεθρο με πολλά είδη θεματικών ε, συνεργασιών. Πλέον μπορούμε να καταγράψουμε τα αποτελέσματα της στρατηγικής αυτής για την ανταλλαγή γνώσεων, την χορήγηση πόρων, την καλύτερη ρύθμιση. Το Κοινοβούλιο, ρωτώ, πώς συμμετέχει, μάλλον πώς ενημερώνεται σε σχέση με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών θα υποβάλλεται εκθέσεις. Πώς θα ενημερώσετε λοιπόν το Κοινοβούλιο που πραγματικά προώθησε και έσπρωξε αυτή την ατζέντα για την Υπέθρο. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να δούμε δηλαδή ποια είναι τα αποτελέσματα και κυρίως σε ό,τι αφορά και την καλύτερη ρύθμιση στο μέλλον για να είμαστε πιο σωστοί στο έργο μας ως συνομοθετής. Ευχαριστώ, σας εύχομαι καλή επιτυχία και στο μέλλον. Θα είναι ένα μέλλον ε, χωρίς την παρουσία μου στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και συμφωνώ με πολλά από τα σχόλια του κ. Φάνιστερ και σας εύχομαι τη καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Όλη την ώρα σκεφτόμαστε την προεκλογική εκστρατεία, ποιος θα είναι εδώ, ποιος όχι. Αλλά αυτό είναι λογικό τέτοια περίεργο εδώ τελευταίες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ρέζη. Κυρία Μάλεβιτς, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και για την παρουσίαση κύριε Λεμέτρ. Αναφερθήκατε στην κατάσταση των πληρωμών ε, για το διάστημα 2014-2020 και το 7-2013 εσείς είπατε ότι είναι καλά. Εγώ δεν βλέπω όμως τίποτα το καλό, διότι το 2020 και το 2025, στο τέλος του πέμπτου έτους ε, εφαρμογής, ε, βλέπουμε τα αποτελέσματα και πάντα καν, το ίδιο, ότι έχουμε καθυστερήσει στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2015 ξεκινήσαμε ε, αμέσως, δηλαδή στην αρχή της νέας περίοδου, να ρωτάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής στα κράτη-μέλη. Αλλά τότε ερχόταν η Επίτροπος εδώ και παρουσίαζε τα μέτρα για την περίοδο 2007-2013. Δηλαδή, κάθε φορά που ξεκινούν οι νέες προοπτικές, ακόμα εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με την προηγούμενη περίοδο και ε, γι' αυτό συνέχεια έχουμε καθυστερήσεις ε, και ελλείψεις στην εφαρμογή στη νέα προγραμματική περίοδο. Τι θα κάνουμε λοιπόν τώρα ώστε να μην επαναλάβουμε τα ίδια σφάλματα στη νέα περίοδο. Ένα από τα μέτρα μας είπατε είναι να ξεκινήσει ο προγραμματισμός στο στομότερο δυνατόν, αλλά όπως ε, ρώτησε και η κυρία Κρέλ, πώς θα γίνει αυτό ε, αφού οι διαπραγματεύσεις για το CPR ε, είναι ακόμα ε, ατελείς και δεν έχουμε συμπεράσματα. Επίσης, στο δικό σας το σχέδιο λέτε ότι μέχρι τέλος Ιουνίου αναμένεται να υποβληθούν ημερομηνίες στόχος για εταιρικέ συμπράξεις και προγράμματα. Και μετά, όταν είδα στην παρουσίαση μέχρι τέλος Ιουνίου, νόμιζα ότι θέλετε αμέσως να λάβετε τα πρώτα σχέδια των ε, ε, συμφωνιών εταιρικής σχέσης ε, από την επόμενη περίοδο. Θα ήταν εξαιρετικό να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να σκεφτούν για προγράμματα στα σκαριά, για συμπράξεις αυτή τη στιγμή, γιατί το 2020 θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία των προγραμμάτων και το 2021 θα περιμένουμε να ξεκινήσουν τα προγράμματα ώστε να μην αντιμετωπίσουμε αντίστοιχα προβλήματα στη νέα προγραμματική περίοδο. Πρέπει να τα επιταχύνουμε όλα. Και αυτά που παρουσιάσετε εσεί είναι πολύ καθυστερημένα. Οι προθεσμίε που μα παρουσιάζετε είναι κατόπιν εορτή. Ξέρω ότι δεν υπάρχει κοινή συμφωνία για το CPR, αλλά όπω είπατε κι εσεί υπάρχουν κάποιε κοινέ θεματικέ προτεραιότητε και γνωρίζουμε κάποια προγράμματα τα οποία θα πρέπει ε, να προχωρήσουν. Ξέρουμε σε ποιους τομείς πρέπει να προετοιμαστούμε και έχουμε πράγματα. Γιατί να μην πιέσουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν για την προετοιμασία προγραμμάτων από τώρα και να μην περιμένουν το 2020. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Νομίζω είναι αρκετές. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερις παρεμβάσεις μεν, αλλά πολύ ψωμί. Πάρα πολλά σχόλια και ερωτήσεις. Πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερως ικανοποιημένος με την ατμόσφαιρα εδώ σήμερα. Είναι κάπως ιδιαίτερη, επιτρέψτε μου να πω. Και καλό θα ήταν να περάσει και στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. οι ανταλλαγές μας έτσι θα γίνουν και πιο ευχάριστες. Κύριε Φανίσερ Ρόι, έχετε απόλυτο δίκιο να τονίζετε το, σύστημα, το πρόγραμμα υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων, το οποίο προτείναμε ως νέο εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να δώσει κίνητρα για έγκαιρες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Χρειάστηκε να αναγνωρίσουμε συλλογικά ότι είναι ανεπαρκής ε, ο δυναμισμός για τις μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώς και θεωρήσαμε ότι πρέπει να υπάρξουν κάποια περαιτέρω κίνητρα θετική φύσεω, να μην είναι κυρώσει, να είναι κάτι θετικό δηλαδή για τα κράτη-μέλη, ώστε να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συστάσεις αναχώρα και να κάνουν κάτι για, για τις συστάσεις. Η μεγάλη διάκριση που θα έκανα όσον αφορά τον καταμερισμό της εργασίας μεταξύ το πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων αφενός και την ε, πολιτική συνοχή και το μέλλον όπως το φανταζόμαστε είναι ότι το πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων δεν θα αφορά συγκεκριμένες επενδύσεις. Όπως γνωρίζετε, πολλές οι μεταρρυθμίσεις είναι θέμα νομοθεσίας και όχι δαπάνικων κονδυλίων. Και θα υπάρχουν ε, οικονομικά κίνητρα απλώς ε, γιατί κάποιος θα αλλάξει τους κανόνες, για παράδειγμα, στα κράτη-μέλα, κανονισμούς για την αγορά εργασίας. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει η πολιτική συνοχή ούτε σήμερα ούτε αύριο, διότι η πολιτική συνοχή αφορά επενδύσεις σε ανθρώπινο και ε, υλικό δυναμικό και είναι πολύ συγκεκριμένε και συνδέονται με συγκεκριμένες δαπάνες ή με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν και εγώ τη μεταφορά σας και θα πω ότι αυτές είναι δύο διαφορετικές πλευρές, όπως τις φανταστήκαμε, του ίδιου νομίσματος και το ίδιο νόμισμα είναι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία είναι χρήσιμα ώστε η Ευρώπη να αναπτυχθεί πιο δυναμικά και σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Ένα επιπλέον σχόλιο επ' αυτού. Όπως γνωρίζετε, στην περίοδο αυτή έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε βάση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και πιο συγκεκριμένα του θεματικού στόχου 11 μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης. και ενίσχυση των διοικητικών δυνατοτήτων. Αυτές είναι οι μορφέ των μεταρρυθμίσεων που στο μέλλον δεν θα χρηματοδοτούνται πλέον στην πολιτική συνοχής, αλλά μπορούν να μεταρρυθμούν, να, ε, χρηματοδοτηθούν μέσω του συστήματος στήριξης μεταρρυθμίσεων. Ε, είναι αλήθεια ότι δεν αναφέρθηκα στο αποθεματικό επιδόσεων και το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα εκεί. Πρόκειται για κάτι το οποίο έχουμε αναλάβει για φέτος. Θα λάβουμε στοιχεία από τα κράτη-μέλη στο τέλος Ιουνίου μέσω των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής και σε αυτές τις εκθέσεις θα μας πούνε ποιο ήταν το αποτέλεσμα για τους διάφορους δείκτες επιδόσεων στο τέλος του 2018. Δεν έχουμε πλήρες πληροφορίες για όλα αυτά ακόμα. Έχουμε κάποια στοιχεία. αλλά ακόμα είναι λίγο εμβαλωματική η εικόνα. Αυτό το οποίο αναμένω είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, δηλαδή δεν θα επιτυγχάνονται οι στόχοι ή το 80% των στόχων στο 1 τρίτο των ε, λεγόμενων ε, δικτών επιδόσεων που σημαίνει ότι θα πάρουμε το αποθεματικό επιδόσεων από κάποιες ε, άξονες προτεραιότητες για να περάσουν σε άξονες προτεραιότητες που έχουν καλύτερες επιδόσεις εντός εισαγωγικών ώστε να συζητηθούν και να αποφασιστούν αυτά με τα κράτη-μέλη. Δηλαδή θα υπάρχουν αλλαγές στα προγράμματα, όταν ε, είναι βέβαια πιο σαφής η εικόνα και όταν έχει κατάλληλη στιγμή. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι είναι μηχανική διαδικασία. Ξέρουμε τους στόχους, είναι ποσοτική και μπορούμε να δούμε εάν πλησιάζουμε το στόχο ή αν έχουμε ξεπεράσει τους στόχους. Αν όχι, οι κανόνες είναι σαφείς. Πρέπει να πάρεις το 6% και το 6% να πάει αλλού. Δεν θέλω τώρα να κάνω εικασίες για το κατά πόσον στο τέλος θα είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ή όχι. Αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι δεν θα περιλαμβάνει και πάρα πολύ στρατηγικό σχεδιασμό. Θα είναι απλώς ε, μετρήσεις βάσει του τρόπου με τον οποίο έχουμε καθορίσει τους στόχους και πολλοί από αυτούς τους στόχους είναι χρηματοπιστωτικοί. Ξοδέψατε τα χρήματα αρκετά γρήγορα. στον τάδε τομέα ή στον δύνατο τομέα. Μπορεί να βρεθούμε λοιπόν ενώπιον τη εξή κατάσταση. Να μην είμαστε πάντα ικανοποιημένοι για το γεγονό ότι κάποιοι τομεί δεν θα μπορούν να υποφοληθούν το αποθεματικού. Θα έχουμε κάποιε περιπτώσει, για παράδειγμα, όπου θα αφαιρούνται χρήματα από ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ε, του κλίματο ε, κλπ. Δεν ε, κάνω πολλέ κασίες, αλλά μπορεί να συμβεί αυτό. Θα πάρουμε τα χρήματα από εκεί και θα τα πάμε σε επιπλέον οδικά ε, έργα. Ε, καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να βρεθούμε ενώπιον τέτοιου διλήμματος. Το κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο, ρωτάει ο κ. Βανίστερ ή απλώς ε, είναι μια διαδικασία που θα είναι κλειστή. Σίγουρα επιθυμούμε να σας ενημερώνουμε πλήρως για τα πορίσματά μας, αλλά και πάλι όλα αυτά γίνονται μηχανικά και μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες. Η διαδικασία είναι τέτοια που δεν επιτρέπει περιθώριο εκτιμήσεων για το κατά πόσον έχεις επιτύχει το στόχο σου ή όχι. Το μόνο στοιχείο επί του οποίου θα υπάρχει περιθώριο για αποφάσεις είναι πού θα πάνε τα χρήματα. Από πού θα τα αφαιρέσουμε είναι σαφές, γίνεται αυτόματα. Αλλά πού θα δοθούν κονδύλια στους τομείς που υποτίθεται έχουν καλύτερες επιδόσεις, εκεί σίγουρα υπάρχει κάποιο περιθώριο επιλογής και επειδή αναφερόμαστε σε επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία τροποποιούνται θα γίνει συνήθως με το κράτος μέλος, θα κάνουμε μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα βλέπουμε από εκεί και πέρα ε, κατά πόσο είναι και δεόντως αιτιολογημένη η πρόταση. Θα ήθελα να κάνω μια σύνδεση με τα όσα έχουμε προτείνει για το μέλλον. Έχουμε προτείνει κάτι άλλο για το μέλλον. Η εικόνα για το πώς θα είναι το ε, αποθεματικό επιδόσεων στην παρούσα περίοδο είναι ο γνώμονας για αυτό το οποίο προτείναμε για το επόμενο διάστημα. Προστείνουμε κάτι πιο έξυπνο για το μέλλον μέσω της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης και της προσέγγισης 5 συν 2. Γιατί εκεί τουλάχιστον δίνουμε πλήρες περιθώριο για νέες αποφάσεις, για νέες προτεραιότητες και δεν συνδέονται αυτές με την εντελώς μηχανική προσέγγιση ε, με την οποία αξιολογούμε τα πράγματα. Χαίρομαι που αναφερθήκατε στα συμφέρον των Υπουργών Οικονομικών, διότι ίσως δεν ήμουν αρκετά σαφής σε αυτό που σας είπα μιλούσα για τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε ότι στο μέλλον δεν θα έχουμε ένα φαινόμενο κατά το οποίο ξαφνικά οι επενδύσεις που υποστηρίζονται στη συνοχή μειώνονται για μια περίοδο μέχρι να αρχίσει σιγά σιγά να λειτουργεί σωστά η νέα περίοδος. Και τόνισα ότι έχουμε προτείνει ένα νέο, πολύ πιο ευέλικτο κανόνα για να επιτρέψουμε κάποια προγράμματα τα οποία ξεκίνησαν σε μια προγραμματική περίοδο να μπορέσουν να συνεχιστούν με χρηματοοικονομική στήριξη αλλά και στην πράξη για την επόμενη περίοδο. Βεβαίως όλα τα χρήματα τα οποία προβλέπονται για το διάστημα 2014-2020 πρέπει να απορροφηθούν στη συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο και δεν μπορούμε να τα προωθήσουμε στο μέλλον. Θέλουμε η χώρα να δαπανά τα κονδύλια της πιο γρήγορα στο μέλλον. Αλλά αυτό θα πρέπει να μας βοηθήσει για να έχουμε μια πιο γρήγορη εικόνα της νέας περίοδου. Γιατί έχουμε κάποια ε, προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται και τα οποία μπορούν ήδη να οδηγήσουν σε επιστροφές ε, πολύ γρήγορα στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Αυτός είναι ένας τρόπος να εξομαλύνουμε λίγο τα πράγματα. Ενώ μέχρι τώρα η αρχή αυτή ότι μπορεί να συνεχιστεί ένα πρόγραμμα στην επόμενη προγραμματική περίοδο ήταν μια πάρα πολύ σπάνια εξαίρεση. Αυτά τα οποία αποκαλούσαμε phased projects. Ε, τώρα πλέον θα είναι πολύ πιο φυσικό να γίνει κάτι τέτοιο και θεωρούμε ότι είναι προς το γενικότερο συμφέρον για να έχουμε ομαλότερες επενδυτικές δραστηριότητες. Και νομίζω ότι αυτό σχετίζεται επίσης και με τα σχόλια της κυρίας Μάλετιτς. Συμφωνώ μαζί σας. Το 2007-2013 δεν ήταν και καμιά περίοδος για την οποία να είμαστε περήφανοι. 25% απλώς τονίζω ότι ήταν τουλάχιστον καλύτερο από εκεί που βρισκόμαστε σήμερα. Και αυτό επαναλαμβάνω, παρά την κρίση του 2009 που ξέρουμε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο ε, διότι πάγωσαν οι επενδύσεις ε, σε όλα τα κράτη-μέλη. Αναφερθήκατε στο 2015 και το γεγονός ότι το 2015 όλοι είχαμε ως στόχο να ολοκληρωθεί το 2007-2013 καλά. Συμφωνώ, ναι. Είχαμε την εξής αιμονή, στο τέλος της περίοδου δεν θέλαμε να έχουμε τεράστιες απώλειες, μέσων βάσει πολιτικής συνοχής, να μείνουν δισεκατομμύρια χωρίς απορρόφηση και δεν, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί όπως πρέπει. Και νομίζω ότι από αυτή την άποψη είχε μεγάλη σημασία να γίνει προσπάθεια γιατί ήταν ουσιαστική η κίνδυνη και τα αποτελέσματα βεβαίως ήταν ενθαρρυντικά γιατί τελικά η περίοδος 2007-2013 θα έχει ένα τελικό ποσοστό απορρόφησης πάνω από το 99% των διαθέσιμων μέσων. Δηλαδή θα είναι πολύ περιορισμένη η έλλειψη δέσμευσης, η, η ακύρωση μιας δέσμευσης. Ε, ελπίζω όμως να μην καθόμαστε συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι απορροφούνται όλα τα χράματα. Επειδή έχουμε χρόνο άπλωτο για το 2014-2020, πολύ περισσότερο από όσο είχαμε περισσότερο, τελικά δεν θα έχουμε αυτή τη δυσκολία απορρόφησης. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ήδη από τώρα στρεφόμαστε με αποφασιστικότητα προς το μέλλον. Και αυτός είναι ο στόχος αυτού που σας παρουσίασα. Να έχουμε ήδη από τώρα, πολύ νωρίτερα από ό,τι στο παρελθόν, μια θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για κάθε κράτος μέλος, δηλαδή ποιες πιστεύουμε εμείς ότι είναι οι προτεραιότητες, να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να σκεφτούν ήδη από τώρα πώς σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τους επόμενους 18 έως 21 μήνες μέχρι το τέλος του 2020 και να πιέσουμε να επιτευχθεί ο κοινός στόχος να εγκρίνουμε συμπράξεις και επιχειρησιακά προγράμματα στο τέλος του 2020 ή αμέσως στην αρχή της επόμενης περίοδου. Αλλά φυσικά εμείς δεν μπορούμε να επαγορεύσουμε στα κράτη-μέλη με ποια ταχύτητα θα δεσμευθούν μαζί μας. Γι' αυτό και σε αυτό το σημείο του ζητάμε απλώς ένα χρονοδιάγραμμα ουσιαστικά, το οποίο θα περιλαμβάνει ως πρώτη ημερομηνία στόχο μια εικόνα για το πότε σκοπεύουν να μοιραστούν μαζί τους ένα πρώτο σχέδιο κειμένου για πρώτες ε, ε, προτάσεις και επιχειρησιακά προγράμματα. Και ελπίζουμε τα κράτη-μέλη να μας δώσουν μια ημερομηνία το συντομότερο δυνατόν και ήδη από φέτος, δηλαδή να μας πούνε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2019 θα σας δώσουμε το πρώτο σχέδιο κειμένου, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να ξεκινήσουμε μάλλον τη συζήτηση πιο συγκεκριμένα. Ρωτήσατε τι άλλα μέτρα λαμβάνονται για να βελτιωθούν οι πιθανότητες η επόμενη περίοδος να ξεκινήσει με μεγαλύτερο δυναμισμό. Πιέζουμε τα κράτη-μέλη επίσης για να επικεντρωθούν στις αδυναμίες τους, στις διοικητικές δυνατότητες που έχουν ήδη από τώρα και μάλιστα προτείναμε οι διαχειριστικές και ελεγκτικές δομές να είναι ίδιες για την επόμενη περίοδο. Επομένω ξέρουν σε ποιε διοικητικέ δομές θα χρειαστούν να επενδύσουν βάσει ε, των αδυναμιών που έχουν αυτή τη στιγμή και εμεί προτείνουμε να επικεντρωθούν σε αυτό από τώρα και θα βοηθήσουμε. Έχουμε ε, προσλάβει και τον ΟΣΑ για να υπάρχει μια σαφή στρατηγική για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις διοικητικές δυνατότητες εκεί που χρειάζεται πριν ξεκινήσει η περίοδος. Και αυτές οι προσπάθειες θα ξεκινήσουν στους επόμενους μήνες. Θα περάσω όμως και σε αυτό το καθόλου θεμητό ερωτηματικό που υπάρχει για αυτή τη φιλοδοξία και την αισιοδοξία ε, που εξέφρασε η κυρία Κρέλ. Συμφωνώ πως αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι για την καλύτερη των περιπτώσεων. Σίγουρα είναι αρκετά φιλόδοξο όμως, σε τελική ανάλυση, η επιτυχία της ε, προσπάθειας αυτής θα εξαρτηθεί από τους εξής δύο παράγοντες. Το κάθε κράτος μέλος, πρώτα, και πόσο φιλόδοξα είναι τα ίδια και πώς θα οργανωθούν για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Αυτό θα φανεί από τον οδικό χάρτη και έπειτα από το ίδιο το χρονοδιάγραμμα όπως είπατε κι εσείς, ε, της επίτευξης συμφωνίας για το ίδιο το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό που είπατε δηλαδή ότι η συμφωνία για το, το ίδιο το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα βασικά του στοιχεία ίσως ε, γίνει πάρα πολύ αργά και ενδεχομένως να καθυστερήσουμε και για το ίδιο το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βέβαια θεωρώ απόλυτα εφικτό να συνεχίσει να σημειώνεται πρόοδος σε αυτές τις διμερείς συζητήσεις για την νομοθεσία, ε, το Ταμείο Συνοχή, το Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη, ESF, ε, ΣΥΝ, κανονισμό περί κοινών διατάξεων κτλ. Παράλληλα με τις συζητήσεις για το πολιτισμο δημοσιονομικό πλαίσιο. Και από όσο γνωρίζω, το Συμβούλιο και το Συνοβούλιο μόλις ε, συμφώνησαν για το InvestEU. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι μπορείς να συμφωνήσεις πάνω σε πολλά θέματα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και σε ό,τι αφορά την ίδια την πολιτική συνοχής, υπάρχουν σε επίπεδο συμβουλίου κάποια θέματα που συνδέονται με το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Όμως οι πρώτοι τριμερείς διάλογοι έχουν δείξει ότι μπορούν να γίνουν πολλά και να βελτιωθούν οι λεπτομερείς ε, διατάξεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε σε μια τελική συμφωνία πολύ σύντομα μετά την έγκριση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Και σίγουρα δεν θα καταφέρουμε να εγκρίνουμε επίσημα τα διάφορα προγράμματα και τις ε, συμφωνίες προτού υπάρχει νομοθεσία. Όμως δεν πρέπει να είμαστε λιγότερο φιλόδοξοι. Αντιθέτως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το διαθέσιμο χρόνο και να καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο. βασιζόμενοι σε αυτές τις εικασίες. Σίγουρα δεν θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε με τα κράτη-μέλη για τις λεπτομέρειες σχετικά με τα νούμερα. Αυτό δεν θα το γνωρίζουμε και δεν θα ξέρουμε ποια θα είναι ακριβώς η πιστώση για κάθε χώρα προτού αυτές ε, δημοσιευθούν. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η θεματική συγκέντρωση ούτε και ποιος θα είναι ο ορισμός ε, του κάθε στόχου πολιτικής. Τις σχετικές ε, δαπάνες που θα υπερβαίνουν τον ε, προϋπολογισμό ή όχι. Δεν ξέρουμε ποια θα, ποιες θα είναι οι εξαιρέσεις για συγκεκριμένες δαπάνες. Αυτό προφανώς χρειάζεται πιο πολύ δουλειά στις λεπτομέρειες έτσι ώστε να γίνει σωστά ο σχεδιασμός, όμως νομίζω πως θα είμαστε πολύ γρήγοροι εάν μέχρι τότε καταφέρουμε να έχουμε σημειώσει πρόοδο για τη στρατηγική, για το μέλλον της ε, συνοχής και των σχετικών δαπανών, για τις προτεραιότητες του κάθε κράτους μέλους και αν έχουμε κάποια ένδειξη της κατανομής των κονδυλίων στα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα και τις διάφορες προτεραιότητες. Ναι, να σας διακόψω λίγο, Πρόεδρος. Ναι, ε, κυρία Κρέλ, δεν το πιστεύω, αλλά τέλος πάντων, πώς θέλετε να ζητήσετε από τα κράτη-μέλη να υποβάλουν προτάσεις για μια συμφωνία εταιρικής σχέσης, ας πούμε, όταν 13 κράτη-μέλη δεν συμφωνούν για την ίδια την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνία εταιρικής σχέσης. Δεν καταφέραμε να συμβαστούμε σε αυτό το θέμα και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο φυσικά θέλουν όλα τα κράτη-μέλη να έχουν υπογράψει τέτοιες συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Τα μισά όμως κράτη είναι υπέρ και τα μισά κατά. Αν ξεκινάμε ήδη με ένα μεγάλο ερωτηματικό, δεν μπορούμε να τελειώσουμε πριν τον Οκτώβριο ή πριν τον Νοέμβριο. Δεν βλέπω λοιπόν ότι έχουμε περιθώρια για συνδοξία. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που αναφερθήκατε σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, διότι συμφωνώ πως αυτή θα είναι και η μεγαλύτερη δοκιμασία για τα κράτη-μέλη. Ε, να δούμε αν έχουν πάρει στα σοβαρά αυτές τις θεσμεύσεις ή όχι. Καταρχάς, ε, δεν πιστεύω πως υπάρχουν 13 κράτη-μέλη που αρνούνται να ε, υπογράψουν συμφωνίες εταιρική σχέσης. Είναι ε, η περίπτωση αυτή διαφορετική. Πρόκειται για εξαιρεσει. Δεν είναι και τα 14 κράτη-μέλη κατά της σύναψης συμφωνίας εταιρικής σχέσης ή έστω μια συμφωνία με αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν επιμέρου ε, διαφωνίε συγκεκριμένα θέματα. Τώρα, γιατί είναι τόσο σημαντική η δοκιμασία, διότι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν βλέπουμε ότι εάν τα στοιχεια υπαρχουν επιμερους διαφωνησεις συγκεκριμενα θεματα τωρα γιατι ειναι τοσο σημαντικη η δοκιμασια διοτι απο την ευρωπαικη επιτροπη εαν βλεπουμε οτι αν τα κρατημελη δεν θέλουν να μας πούν ποιοι ακριβώ είναι οι στόχοι στρατηγικής για την πολιτική συνοχή στο μέλλον, δεν πρόκειται να γίνει καμία συζήτηση. Και δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε συζητήσεις για κάποια αόριστα και προγράμματα. Χρειάζεται συγκεκριμένη λεπτομερής προσέγγιση από το κάθε κράτος μέλος. Και δεν λέμε πως σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να έχουμε όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές, ας σκεφτούμε πρακτικά και πρέπει επιτέλους, αν ε, το κάνουμε αυτό, να δούμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν συμφέρον να συνεργαστούν μαζί μας. Και δεν θέλω να κατονομάσω κράτη-μέλη, όμως ε, υπάρχουν κάποια τα οποία στηρίζουν αρκετά περίεργα, στο πούμε έτσι, προγράμματα. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν δεν θα έλεγα πως είμαι απεσιόδοξος γιατί στηρίζομαι στην ικανότητα των κρατών μελών να αναγνωρίσουν το γεγονό ότι πρέπει να μιλήσουμε επί τη ουσία, πρέπει να μιλήσουμε για αυτά που είχαμε προτείνει στι συμφωνίε εταιρικέ σχέσει. Διαφορετικά, αυτέ οι διμερεί συζητήσει δεν θα σημειώσουν καμία πρόοδο. Κύριε Βαν Μίλτενπουργκ, σωστά καταλάβατε ότι εμέσω πρότεινα να επιστρέψουμε στον ίσινδιο, Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι προτείναμε και μια προοδευτική επιστροφή σε αυτό τον ίσινδιο και όχι ε, μια επιστροφή με τρόπο που θα είναι που θα έχει δυσάρεστες συνέπειες. Θα αναπότομος. Βέβαια το πώς θα επιστρέψουμε στον ΙΣΙΝ 2 είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε. Τώρα για τις μεταφορές από το ΣΕΦ, συνδέοντας στην Ευρώπη. Θα είμαι ειλικρινής, όσο μπορώ. η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επαναληφθούν αυτές οι μεταφορές σε αυτή την περίοδο είναι κάτι που θεωρούμε θετικό, κάτι που έχει ισχυρές βάσεις και θα οδηγήσει θετικά αποτελέσματα. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακόμα με βεβαιότητα αν οι φάκελοι των κρατών μελών που έχουν μεταφερθεί θα ε, τηρηθούν στο 100% από το κάθε κράτος μέλος. Θα υπάρχουν κάποια, κάποια κράτη που θα κερδίσουν, κάποια κράτη που θα χάσουν. Αυτό βέβαια θα το δούμε και στο μέλλον και θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή και την υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν επιλεγεί. Για μας αυτό ήταν πάντα στο παιχνίδι, διότι είχαμε συμφωνήσει να προστατεύονται οι εθνικοί φάκελοι μόνο για τα πρώτα τέσσερα χρόνια του τρέχοντος πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Δεν θεωρούμε λοιπόν πως είναι προβληματική η ανακατανομή έτσι, σε μικρή κλίμακα ή πως έχει αποτύχει το πρόγραμμα και σίγουρα η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της Κομισιόν ήταν πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι στο τέλος θα γίνουν σεβαστοί οι αρχικοί εθνικοί φάκελοι και θα επιτευχθεί η κατάλληλη εφαρμογή και υλοποίηση των επιλεγμένων προγραμμάτων. Τώρα, ε, για τις μη επιλέξιμες δραστηριότητες. Να πω καταρχάς πως χαίρομαι πάρα πολύ που το αναφέρατε, διότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την κατεύθυνση που έχει επιλέξει η συγκήτρια και μάλιστα ανησυχούμε αρκετά, θα έλεγα. Θεωρούμε λοιπόν ότι η προσέγγιση αυτή μας πηγαίνει προς τα πίσω και όχι προς τα εμπρός. Είναι υπέρ το δέον συντηρητική και χαλαρή στην χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αναφερθήκατε σε κάποιους τομείς που θεωρείτε πως θα πρέπει να γίνουν επιλέξιμοι. Ε, θα μπορούσα να προσθέσω κι εγώ άλλον έναν. Για να αιτιολογήσω αυτήν την ανησυχία μας. Οι μέχρι και οι χωματερές θα μπορούν να είναι επιλέξιμες στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε την εξή ερώτηση. Θέλουμε η, η πολιτική συνοχής να εναρμονιστεί πλήρως με την πιο θεμελιώδη βασική στρατηγική που σχεδιάζουμε. για μένα δεν πρέπει να μείνουμε πίσω στην καινοτομία, στην έξυπνη Ευρώπη όπως λέμε. Και δεύτερον, θέλουμε μια πράσινη Ευρώπη, μια βιώσιμη Ευρώπη που να προστατεύει το κλίμα, να καταπολεμήσει τη χρήση, να λόγει τη χρήση πλαστικού, να επιτύχει τους στόχους για το κλίμα κτλ. Τώρα, η πολιτική συνοχής δέχεται μεγάλες πιέσεις οικονομικά. Ας δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το πολίτεσμο συνομικό πλαίσιο, αλλά θεωρώ πως δεδομένων όλων αυτών των ε, στοιχείων που δίνουν βεβαιότητα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί προ ε, τι θέλουμε να περιέχει πολιτική συνοχής και τι συμφωνίε συνάπτουμε. Χρειάζεται συνέπεια λοιπόν με τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται να είμαστε πιο επιλεκτικοί από ό,τι στο παρελθόν. Γι' αυτό και επιμένουμε στο ότι δεν θα πρέπει στο μέλλον να χρηματοδοτούνται τεχνολογίες που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα, ε, στο, στα περιφερειακά αεροδρόμια, για παράδειγμα, στις ε, χωματερές, όπως είπα, κτλ. κτλ, κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο λοιπόν της όλης συζήτησης, διότι αυτό θα καθορίσει εν μέρη και την εικόνα της πολιτικής συνοχής. Να κάνω ένα σχόλιο. Αναφερθήκατε στις κάτω χώρες και τις δαπάνες, στα καινοτομία κτλ. Αν όμως συγχωνευτεί το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με το Ταμείο Συνοχής, τότε η μετάβαση, για παράδειγμα, από τα ορυκτά καύσιμα σε πιο βιώσιμα καύσιμα δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, θέλει χρόνο. Εσείς θα στηρίζετε λοιπόν επενδύσεις σε αυτό, σε αυτή τη μετάβαση ή όχι. Επίσης, πολλά προγράμματα του Ταμείου Συνοχής βασίζονται, ε, μάλλον πολλά προγράμματα έχουν να κάνουν με τα απόβλητα, διαχείριση απορριμμάτων κτλ. Στις χώρες της συνοχής όμως υπάρχουν μεγάλα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν. Για παράδειγμα, όπου γίνεται όπου υπάρχουν χωματερές, πρέπει να φεύγουν τα νερά που συγκεντρώνονται εκεί. Βλέπετε λοιπόν ότι συνδέονται μεταξύ τους όλα αυτά και χρειάζεται να κάνουμε συμβιβασμούς διότι είναι απαραίτητο. Επιτρέψτε μου να μιλήσω για αυτή την ε, πεποίθηση ότι το πρόβλημα μπορεί να είναι το RDF και ο κανονισμό μαζί. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί, θεωρώ. Το πρόβλημα είναι η πολιτική επιλογή, πολιτικές επιλογές που κάνουμε εμεί. Γιατί η χρηματοδότηση που επιτρέπεται από τα Ταμεία συνοχή είναι εξίσου δυνατή και στα πλαίσια του RDF. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι τι είδους περιβαλλοντικά προγράμματα σε ό,τι αφορά το Ταμείο Συνοχής θέλουμε να υποστηρίξουμε. Και πάλι πιστεύω ότι το σημείο εκκίνησης θα πρέπει να είναι τι είδου στόχου έχουμε θέσει Για τα απορρίμματα, για παράδειγμα, έχουμε πει ότι μέχρι το 2035 θα πρέπει να έχουμε μόνο 10% τέτοιων ε, απορριμμάτων στις χωματερές. Σήμερα απέχουμε πάρα πολύ από το στόχο αυτό και έχουμε ικανότητες στις χωματερές οι οποίες είναι εντελώς ε, δυσανάλογες σε σχέση με αυτό. Τώρα θα επιτρέψουμε να δαπανώνται πόροι για τις κομματερές, για μένα δεν έχει νόημα, δεν στέκει, δεν συνάδει με τον στόχο μείωσης των ικανοτήτων ε, και των, της χωρητικότητας των χωματερών. Σύμφωνα με τους ποσοτικοποιημένους στόχους. Είναι ένα από τα σημεία τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη Και σε ό,τι αφορά την ε, καύση των απορριμμάτων. τα οποία, την οποία θέλουν κάποια κρατημέλη να επιτραπεί για την επόμενη περίοδο. Κοιτώντα του στόχου ε, ανακύκλωση για το 2030-2035, αυτό τι σημαίνει ότι σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση θα έχουμε τεράστιες ε, δυνατότητες και ικανότητες για τέτοιες μονάδες αποτέφρωσης απορριμμάτων. Έχει νόημα λοιπόν να γίνουν δαπάνες. Δεν θέλω να επεκταθώ σήμερα. Και ελπίζουμε τελικά να καταλήξουμε σε κάποιον σωστό συμβιβασμό. Και εγώ ευχαρίστω να δεσμευτώ και να υποσχεθώ στην Επιτροπή Περιφερειακή ανάπτυξη. ακόμα και αν εσεί, ε, κύριε Εμφανίλη, δεν πρόκειται εδώ πέρα την επόμενη περίοδο σε θέματα ε, ατζέντα για την ε, Ήπεθρο και σε ό,τι αφορά τις θεματικές ενότητες που υπάγονται σε αυτή την ατζέντα. Αυτά. Και το ίδιο θα μπορούσα να πω και προς τον κύριο Φανίστελ για τις προπαρασκευαστικές τράσεις μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Ξέρετε, Εγώ ευχαρίστω να σας δώσω την αξιολογήσή μας για το πού βρισκόμαστε. Μάλιστα. Μία άλλη ερώτηση. Ο στόχος αυτός μέχρι το 2029, μέχρι το 2030 να έχουμε μία ποσόστοση η οποία εξ αρχής ήταν μία ρεαλιστική. Δεν είναι πρώτη φορά, ξέρετε, που συμβαίνει κάτι τέτοιο, να θέτουμε έναν ρεαλιστικό στόχο και από ό,τι προκύπτει και η Γερμανία και η χώρα μου δηλαδή παρουσιάζει την κύκλικη οικονομία, αλλά είναι η χώρα που στέλνει τα σκουπίδια της, τα πλαστικά της δηλαδή κυρίως στην Ασία. Και τώρα έρχεται η Μαλαισία και λέει ότι κοιτάξτε δεν τα χρειαζόμαστε τα σκουπίδια σας. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα για ένα μεταβατικό στάδιο να μην γίνεται αποτέφρωση έχει, υπάρχουν καλές τεχνολογίες, πολύ καλές τεχνολογίες waste to energy για το πώς μπορούμε να παράγουμε ενέργεια από τα σκουπίδια, από την αποτέφρωση πλαστικών όλος ιδιαίτερος. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια δυνατότητα προκειμένου χώρες οι οποίες δεν μπορούν να κάνουν τη δικασία αυτή με δικό του κόστος γιατί είναι πολύ ακριβό να έχουν την ευκαιρία με την πολιτική συνοχή, με τα περιφερειακά μάλλον μέσα, να υλοποιήσουν τέτοιες λύσεις. Τουλάχιστον ε, προσωρινά για την αντιμετώπιση του προβλήματος ε, και για να παράγουμε και ενέργεια. Να μην υπάρχει τόσο αυστηρή οριοθέτηση λοιπόν, γιατί έτσι και αλλιώς τους στόχους ε, για, που είχαμε θέσει δεν πρόκειται να το πετύχουμε. Το ξέραμε αυτό αυτή τη αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρο. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Σύμφωνο, συμφωνώ ότι θα πρέπει να ζητήσουμε εύλογου ε, συμβιβασμού. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι σε αυτού του συμβιβασμού, σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να αμελήσουμε του στόχου που έχουμε θέσει. Τώρα ποιο είμαι εγώ να, να κρίνω αν είναι ρεαλιστική ή όχι η στόχη αυτή για το 2025. Εγώ απλά σημειώνω ότι έχει αποφασίσει ο νομοθέτης, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και είναι στόχοι συγκεκριμένοι αυτοί σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα. Να προτείνω ότι ναι, συμφωνώ με τα διάφορα στοιχεία τα οποία έθεσε ο κύριος Τσέλερ, αλλά η τεχνολογία αυτή είναι εξαιρετικά ακριβή. Άρα δεν είναι αυτή μια επένδυση για 5-10 χρόνια αυτό θα μείνει μαζί μας σε μεγάλο βαθμό χρόνου και στην περίπτωση αυτή ενδεχομένως να καταστεί εξαιρετικά μη αποδοτικότητα με εξαιρετικά υψηλό κόστος ε, συντήρησης και η νομοθεσία δεν θα υποστηρίζει για πάντα τη συντήρηση των ε, εγκαταστάσεων αυτών. Μια και λοιπόν αυτή η όθηση για τέτοιου είδους επενδύσεις προέκυψε κυρίως από την περιοχή της Βαλτικής. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή τι είδους κίνητρα δίνουμε. Και κατά πόσο δημιουργούμε ένα πλεόνασμα ικανοτήτων τέτοιων δηλαδή, Έχουμε τρεις τέτοιους αποταυτήρες στη Βαλτική σήμερα. Αν ε, πάρουμε στα σοβαρά τους στόχους που έχουμε θέσει για την ανακύκλωση, αν πάρουμε υπόψη το γεγονός ότι αυτές οι χώρες ε, δημογραφικά μειώνονται ως προς τον πληθυσμό τους. Ε, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου οι δύο τεράστιοι αυτοί αποτεφρωτήρες θα καλύπτουν σε κάθε περίπτωση πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα από τις ε, ανάγκες αποτέφρωσης των τριών βαλτικών χωρών. Άρα, θέλουμε άλλον έναν από το βραδυρά στη Βαλτική. Ναι ή όχι. Και κάτι άλλο που πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σχετικό για, τα, για τις χώρες της Βαλτικής. Οι χώρες της Βαλτικής σήμερα έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά ανακύκλωση κάτω από το 25%. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι 75%. Άρα, τι είδου κίνητρα χορηγούμε αν ε, χρηματοδοτήσουμε από τεφρωτήρες ε, ε, απορριμμάτων που αποτελούν ουσιαστικά την εύκολη λύση για να αποφύγουμε την ανακύκλωση. Ε, όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε ένα κάποιον συμβιβασμό. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση και πραγματικά τη χρειαζόμασταν αυτή τη συζήτηση. Μετά από τόσες συζητήσεις που έχουμε κάνει για τους κανονισμούς κοινωνικών διατάξεων, είναι σαφείς οι διαφορετικές απόψεις επί του θέματος πλέον. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ αισιόδοξη ε, προσέγγιση σας για την ε, προγραμματισμό για την επόμενη περίοδο. Σας ευχόμαστε και κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας. Και εδώ ολοκληρώθηκε η ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος έχει να υποβάλει κάτι υπό τα διάφορα. Όχι. Να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα είναι και η τελευταία στην τρέχουσα θετία. Τη Επιτροπή ε, Περιφερειακή Ανάπτυξη. θα λάβει η χώρα εδώ στις Βρυξέλλες στις 11 Απριλίου από τις 10 το πρωί. Να ευχαριστήσω τους Γερμινείς, λέει η και εμεί σας ευχαριστούμε και πέρα στη συνεδρίαση ε, για σήμερα.